Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε, δεν κατάλαβα τι έγινε με την ψηφοφορία. Ψηφίσαμε για την ημερήσια διάταξη που αποφασίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων ή κατά. Κατά. Ε, Οπότε δεν θα συνεδριάσουμε την Πέμπτη. θέλετε να πληρωθείτε χωρίς να ψηφίσετε. Κύριε Πρόεδρε Ντόλ, κύριε Ντόλ, Ζωζεφ, ψηφίσαμε για ένα μόνο πράγμα. Την Πέμπτη δεν θα γίνει ψηφοφορία για μία μόνο έκθεση, μία μόνο έκθεση δεν θα ψηφίσουμε για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη λαοκρατική δημοκρατία του Κονγκό. Θα συζητήσουμε όλα τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δεν αλλάζουν, αλλά δεν θα γίνει ψηφοφορία για αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση. Ψηφίσαμε μόνο για αυτή την έκθεση. Όλα τα άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη και όλες οι άλλες ψηφοφορίες δεν αλλάζουν. Υπήρξα σαφής. έχουμε μιλήσει, μιλήσαμε μόνο για μια ψηφοφορία. Αυτή την Πέμπτη θα εργαστούμε κανονικά. Είναι σαφές, έγινα κατανοητός. Συνάδελφοι, μιλούσαμε για μία μόνο ψηφοφορία. Μόνο Η συζήτηση αφορούσε μόνο μία ψηφοφορία την Πέμπτη. Για το Κονγκό για την περίπτωση του Κονγκό, της λαοκρατικής δημοκρατίας του Κονγκό. Για τίποτα άλλο δεν μιλούσαμε, μόνο για αυτή την ψηφοφορία. Οπότε, τώρα αρχίζει η συζήτηση. Θα εξετάσουμε την έκθεση της κυρίας Κριστίν Ντεβεράκ, διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. Δίνω το λόγο στην κυρία Ντεβεράκ την εισηγήτρια. Έχετε το λόγο κυρία Ντεβεράκ. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών δεν αφορά μόνο οικονομικούς στόχους, αλλά κυρίως ε, εκφράζει τη βούληση να τηρηθούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την προστασία των ταξιδιωτών. everything is ready. Μπορείτε να συνεχίσετε. Αυτό είναι ένα στόχο τον οποίο πλησιάσαμε, προσεγγίσαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειε μα για να εξασφαλίσουμε βέλτιστο ε, βαθμό ε, ασφάλεια για τι αεροπορικέ μετακινήσει. Γι' αυτό προ, προ, καταθέσαμε αυτή την έκθεση για τη διερεύνηση και πρόληψη των αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. Μετά από δύσκολε διαπραγματεύσει, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού καταφέραμε να βρούμε μια λύση στην πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο που εγγυάται σημαντικές προόδους σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση και πρόληψη των αεροπορικών και τη φροντίδα των οικογενειών των θυμάτων. Εάν επιβεβαιωθεί από την αυρενή ψηφοφορία αυτό σημαίνει ότι τα τέλος του 2010 τα μέτρα που προβλέπουν σε αυτό το κείμενο θα αρχίσουν πλέον να ισχύουν. Ποια είναι τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτή την έκθεση. Πρώτα, ο κανονισμός ενισχύει την ανεξαρτησία. Με συγχωρείτε κυρία Ντεβεράκ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι. Υπάρχει πολλή φασαρία στην αίθουσα. Yes, madam. Please, madam, please continue. Κύριε Ντεβεράκ, μπορείτε παρακαλώ να συνεχίσετε. Λοιπόν, ποια είναι τα μέτρα που προβλέπει αυτή η έκθεση. Πρώτον, την ανεξαρτησία της ε, διερεύνησης και των ερευνητών οι οποίοι θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα αναγκαία μέσα για να προσδιορίσουν τα αίτια του ατυχήματο. Δεύτερο σημαντικό σημείο, η έκθεση αυτή μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε το ρόλο της ΆΙΣΑ σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματο. Προβλέπει σαφώ ότι η υπηρεσία ενεργεί ω αρχή πιστοποίηση. Βλέπω ότι το θέμα δεν φαίνεται να μην ενδιαφέρει κανέναν. Δεν μπορώ να ακούσω ούτε τη δική μου τη φωνή, οπότε να σταματήσω. Μπορείτε παρακαλώ να συνεχίσετε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη διαδικασία. Δεύτερο σημαντικό σημείο. Διευκρινίζει το κείμενο το ρόλο της Άιζα σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος. Προβλέπει ότι ενεργεί ως αρχή πιστοποίησης διερευνά διότι ε, χωρίς να διερευνήσει τα αίτια των ατυχημάτων, αλλά έχει πρόσβαση σε αναγκαία στοιχεία για λόγους πιστοποίησης και μπορεί επίσης να συνδράμει με την εμπειρία της τους ερευνητές. Το κανονισμός προβλέπει ότι σύμφωνα με το παράδειγμα 13 της Σύμβασης του Σικάγο, η ΆΙΣΑΣ θα συμμετέχει στις έρευνες ως, υπό την ιδιότητα του Συμβούλου τρίτη πρόοδος του κανονισμού, η δημιουργία ενός δικτύου ε, αρχών διερεύνησης και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η συνεργασία που ήδη υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών ενώ ε, υπάρχει, θα έχει μία ε, ευέλικτη δομή χωρίς νομική μορφή αυτό το δίκτυο συμβάλλοντας στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών την ανταλλαγή και ε, των βέλτιστων πρακτικών και την κατάρτιση των ερευνητών επίσης των ανακριτών. Επίσης δημιουργεί μια σχέση ανάμεσα στην νομική και την τεχνική έρευνα για τα θέματα ασφάλειας. Ο κανονισμός σημειώνει ουσιαστικές προόδους παρόλο τα, τα διαφορετικά νομικά συστήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Εγγυόμενος μια άμεση πρόσβαση των ανακριτών στα αποδεικτικά στοιχεία και προβλέποντας μια προκατακτική συμφωνία ανάμεσα στις νομικές υπηρεσίες και τις ανακριτικές αρχές. Κάτι άλλο σημαντικό, η προστασία των και των οικογενειών τους. Το κείμενο προβλέπει σε περίπτωση ατυχήματο, ο κατάλογος των επιβατών στο αεροσκάφο ε, ε, που υπέστη ατύχημα πρέπει να είναι διαθέσιμος το αργότερο μέσα σε δύο ώρες, ώστε να μειωθεί η οδυνηρή αναμονή των μελών τη οικογένεια. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης μια σειρά από μέτρα που αφορούν τι οικογένειε των θυμάτων, δυνατότητα τη στιγμή της κράτησης να αναφέρει εν, κάποιος ένα άτομο επαφής μετά από ατύχημα, να ενημερώνει την οικογένεια την πρόοδο της ανάκρισης και των ερευνών, η εμπιστευτικότητα σε ό,τι αφορά την παρουσία στο αεροσκάφος κάποιου ατόμου, αν το ζητήσει η οικογένεια, η επιλογή ε, συγκεκριμένων ατόμων που θα ε, ενεργούν ο σύνδεσμος ανάμεσα στις υπηρεσίες, στις αρχές και τα, μέλη της οικογένειας των θυμάτων, η υποχρέωση για όλες τις αεροπορικές εταιρείε στην Ευρώπη να έχουν ένα σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης που θα προβλέπει και ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων και η δυνατότητα ε, να υπάρχει μια ελάχιστη ασφάλεια αποζημίωσης των θυμάτων. Άλλο σημείο σημαντικό του κανονισμού είναι η αναφορά για τα περιστατικά. Σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την πρόληψη των ατυχημάτων. Εφόσον το κείμενο προβλέπει ότι η ΆΙΣΑ και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων για τα αεροπορικά ατυχήματα. Αυτή η βάση δεδομένων θα αναλυθεί ώστε προληπτικά μέτρα να μπορούν να λαμβάνονται ώστε να αποφεύγεται με τον τρόπο αυτό η να προκύπτουν ατυχήματα. Αυτό είναι το αποτελέσμα του συμβιβασμού. Ευχαριστώ τους σκιώδει εισηγητές με του οποίου είχαμε θαυμάσια συνεργασία και που μα επέτρεψαν, επέτρεψαν να φτάσουμε σε αυτό το ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντεβεράκ. Εγώ δεν σας ε, ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κάνετε γιατί μετά από ξεκινήσατε την ομιλία σας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες στην αρχή. Point of order. Yes, please. Ε, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα πιο πριν να αναφερθώ και δεν ήθελα να διακόψω την εισηγητρία. Σας δίνω απόλυτο δίκιο. Είναι απαράδεκτο Πώ έγιναν τα πράγματα στην αρχή, στην έναρξη αυτή τη συζήτηση. Σε αυτή τη συζήτηση πρόκειται για ατυχήματα αεροπορικά, για ανθρώπινε ζωέ, για πράγματα δηλαδή που αλλάζουν και πώ μπορούν να αλλάζουν την ανθρώπινη ζωή και πώ η ανθρώπινη ζωή μπορεί να προστατευτεί. Είναι σοβαρό το θέμα και θα έπρεπε στο μέλλον να αποφεύγουμε τέτοιο χάο στην έναρξη μια συζήτηση, ιδίω όταν πρόκειται για τόσο σοβαρά θέματα. Ευχαριστώ. Uh, Σα ευχαριστούμε πολύ είναι ένα ζήτημα το οποίο τίθεται σε σχέση με όλους τους συναδέλφους. Είναι πολύ σημαντικό όλοι να μπορούν να αναχωρήσουν το δυνατόν νωρίτερα από την αίθουσα ώστε να παραμείνουν όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση και οι συζητήσεις να γίνονται εκτός αιθούσης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας συνάδελφε. Σας ευχαριστώ. Εξώματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Επίτροπος κυρία Σεσίλια Μάνστρομ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον λόγο κύριε Μάνστρομ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, καλό σας απόγευμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Ντεβεράκ, και τους σκιώδεις εισηγητές επίσης για την προσπάθεια την οποία έκαναν και για την υποστήριξη την οποία έδωσαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτόν τον νέο κανονισμό που αφορά την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ευρώπη. Δεν ήταν εύκολο το θέμα όπως είπε και η κυρία Ντεβεράκ. Αντίθετα περιλαμβάνει θέματα τα οποία είχαν απαιτήσει πολύ ευαίσθητες διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα για την ασφάλεια και στις απαιτήσεις των αρχών της δικαιοσύνης κτλ να διασφαλίσουμε και τις ανακριτικές διαδικασίες όπως επίσης και την ανωνυμία αυτών οι οποίοι θίγονται από τις έρευνες αυτές. Πάντως προχωρήσαμε γιατί θέλουμε να υπάρχει σωστό αποτέλεσμα και να ρυθμίσουμε κάποιους κανόνες οι οποίοι να είναι αποτελεσματικοί, επαγγελματικοί και να αποτρέψουν στο μέλλον πιθανώς κάποια ατυχήματα και να διασφαλίσουν υψηλά επίπεδα ασφαλείας για τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν και για το Συμβούλιο και για το Κοινοβούλιο ε, που προχώρησαν στις απαιτούμενες ε, ε, μορφές συνένεσης. Εμείς συμμεριζόμεθα σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή της αντιλήψης της εισηγητρίας. Νομίζουμε ότι το πράσινο βιβλίο είναι κάτι το οποίο δείχνει ε, ότι χαρακτηρίζεται από μια ε, ισορροπημένη θα έλεγα αντιμετώπιση των προβλημάτων. Βασικός μας στόχος είναι η ασφάλεια των επιβατών. Είναι η βασική μας προτεραιότητα και ήταν πάντα η βασική μας ανησυχία στα πλαίσια των συζητήσεων μέχρι τώρα. Θα ήθελα να προσκαλέσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπερασπιστούν και να εγκρίνουν τελικά την προτινόμενη συμβιβαστική πρόταση. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πίτροπε. Και τώρα εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ακούσουμε τον κύριο Βέρνερ Κούν. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε Μάμστρομ, αγαπητοί συνάδελφοι. Η συνάδελφη, συνάδελφος μας Κριστίν Τεβεράκ συνέταξε μια εξαιρετική έκθεση που μας παρουσίασε μετά από μακρότατες διαπραγματεύσεις. Αλλά προηγούμενα σωστά αναφέρθηκε εισαγωγικά ότι εδώ πρόκειται για ανθρώπινες ζωές και πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε απλά τι γίνεται σε σχέση με την εξέταση αυτών των ατυχημάτων και τώρα πώς σε σχέση με μια οδηγία του 1994 στην οποία αναφερόμαστε, δηλαδή εντωμεταξύ έχουμε μια κοινή αγορά εναέριων μεταφορών. Έχουμε το European Open Sky, τους ανοιχτούς εθέρες. Οι αεναρίες μεταφορές κατά τα τελευταία 15 χρόνια υπερδιπλασιάστηκαν στην Ευρώπη. Οι κοινέ μας προσπάθειες στοχεύουν φυσικά οι ασφάλειες εναέριες μεταφορές να βελτιώνεται διαρκώς. Και είναι απόλυτα επιτακτική ανάγκη όλα τα συμβάντα και όλα τα ατυχήματα σε βάθος να εξετάζονται με κάθε λεπτομέρεια. Και αυτό αναφέρθηκε και από την συνάδελφο Ντεβεράκ και από το πεδίο έντασης που δημιουργείται μεταξύ των δικαστικών αρχών και των ανεξάρτητων ανακριτικών αρχών. Και στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Αερομεταφορών θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και πρέπει να την ενισχύσουμε σε σχέση με αυτό, αλλά και οι εθνικές αρμοδιότητες που υπάρχουν πρέπει ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα, όπως το έχουμε και με την Ομοσπονδιακή Αρχή Εναέριων Μεταφορών στη Γερμανία, να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες ώστε σε βάθος και με απόλυτη ακρίβεια να αναλύονται τα δεδομένα ώστε να μπορούμε να δούμε τι γίνεται με τα σωστά πορίσματα και έτσι να μην διασπαθίζονται κονδύλια σε σχέση με νέε υπηρεσίε και νέου οργανισμού και να υπάρξει εξοικονόμηση κονδυλίων και να συνεργαζόμαστε πιο αποτελεσματικά έτσι μεταξύ μα. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενο ε, ομιλητή είναι ο κύριο Μπράιν Σίμψον, εξ ονόματο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη σκληρή δουλειά που έκανε για το σημαντικό αυτό θέμα και θα ήθελα να εστιαστώ σε δύο θέματα που αναφέρονται στην έκθεση. Πώς πρώτον μπορούμε να βελτιώσουμε την διερεύνηση ατυχημάτων και δεύτερο θέμα τα δικαιώματα των θυμάτων και των συγγενών και των μελών των οικογενειών. Η Επιτροπή Μεταφορών έχει ενισχύσει τις διατάξεις που είχε αρχικά προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσδιορίσαμε το ρόλο της ΕΑΣΕ, όπως είπε η συγγήτριά μας, σε ό,τι αφορά την διερεύνηση ατυχημάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι διερευνήσεις αυτές γίνονται με τελείως αντικειμενικό τρόπο, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Δεν μπορεί η ρυθμιστική αρχή να είναι παράλληλα και ανακριτής. Σε ό,τι αφορά τον σαφή ορισμό του ρόλου της ΕΑΣΕ ως ε, ε, συμβούλου. Αυτό ορίζεται στο άρθρο 14 του ΑΕΚΑΟ. Επίσης πρέπει να προσδιοριστούν ποιες θα είναι οι διερευνητικές αρχές και ποια θα είναι τα στοιχεία τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε την ανάγκη για ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων και αναφορών και ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών που προκύπτουν από ατυχήματα και συμβάντα και όπως επίσης να φροντίσουμε για κατάλληλη αποζημίωση για τα θύματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια ευκαιρία να ξαναδεί το θέμα της προστασίας των, θυμάτων, των δικαιωμάτων των θυμάτων και των συγγενών επιμένοντας να υπάρχει βοήθεια και ενημέρωση σε, σε διάστημα διάστημα δύο ώρων. Πρόεδρε, θέλουμε να πούμε στην Επιτροπή ότι είναι σημαντικό η, οδηγία, η τρέχουσα οδηγία να αναθεωρηθεί ώστε και οι δύο να αλληλοσυμπληρώνονται. Πρόεδρε, νομίζω ότι πρόκειται για πάρα πολύ καλή δουλειά και θέλω να συγχαρώ ακόμα μια φορά του εισηγητέ και τους και εισηγητέ για τι προσπάθειέ του. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σα, αγαπητέ συνάδελφοι και ότι τηρήσατε το χρόνο σα, Ο κύριος Γίλκο Κάτσιν. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρία Μάλμστρομ, αγαπητοί συνάδελφοι. Με μεγάλη περηφάνεια έχουμε αυτό το έγγραφο μπροστά μας, το οποίο α, είναι αποτέλεσμα επιτυχών τριμερών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για τα επιτεύγματά της, για το θάρρος της. Δημιουργήθηκε έτσι ένα πλαίσιο το οποίο οδηγεί σε πολλά ωφέλη και πλεονεκτήματα για τους επιβάτες και το κοινό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα. Η Επιτροπή Μεταφορών προετοίμασε ένα καλό έγγραφο κατά την προηγούμενη άνοιξη, που ήταν και η βάση για τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης ε, την Ένωση των Ελεγκτών Εναερίων Μεταφορών, που και αυτή συμμετείχε στην προετοιμασία αυτής της πρότασης. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορέσαμε να έχουμε την, ε, να αντιμετωπίσουμε το θέμα των αλλαγών του ρυθμιστικού πλαισίου ή των ε, διατάξεων κατά την επεξεργασία. Θα ήθελα να πω ότι απόλυτη ελευθερία έρευνα θα έπρεπε να δίνεται στους ε, ερευνητές. Δεν θα έπρεπε να γίνονται τα πράγματα βιαστικά ο ρόλος των δικαστικών αρχών και των ανακριτικών αρχών θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια και έτσι να δρούμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι οι τεχνικές ε, εξετάσεις θα πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε ανάμειξη από πλευράς των δικαστικών αρχών ή των δικαστών. Θα πρέπει να αποφύγουμε οποιασδήποτε αναμίξεις και όλα τα ατυχήματα και συμβάντα, όχι μόνο εκείνα τα οποία οδηγούν σε μια τραγική έκβαση και οτιδήποτε αντιβαίνει την ασφάλεια θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να αντιμετωπίζεται και σε σχέση με την ε, οδηγία αυτή θα πρέπει να αναδιατυπωθεί το δυνατόν ε, ταχύτερα. Η ΑΙΑΣΑ έχει αναλάβει ένα σαφέστατο ρόλο, δεν είναι ε, ερευνητική αρχή, έχει συμβουλευτικό ρόλο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας και μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές. Η ερευνήτρια έλαβε υπόψη τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία προτείναμε και ευχαριστώ. Μπεργα στην συνέχεια, παρακαλώ, εξ ονόματος των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η έκθεση στη σημασία της ε, δεν μπορεί να ε, ε, υπερεκτιμηθεί, διότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο δίνει τις πληροφορίες εκείνες συνολικά που στο παρελθόν ήταν κατακερματισμένες και δεν μπορούσαν να είναι σφαιρικές και δεν ήταν δικτυωμένες. Σε ένα, ε, μια χρονική περίοδο τεράστιας ε, πίεσης από τον ανταγωνισμό στις ενέργειες μεταφορές είναι αναγκαίο, είναι επιτακτική ανάγκη εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα να μπορούν να προστατεύονται από την άσκηση πίεσης από ανταγωνίστριες ε, αεροπορικές εταιρείες και άλλους ανταγωνιστές. Εδώ πρέπει να μεριμνήσουμε αυτές στις τις πληροφορίες που τις χρειαζόμαστε επιτακτικά για την πρόληψη, να μπορέσουμε να τις προστατέψουμε και να προστατέψουμε αυτούς τους ανθρώπους και να υπάρχει μια ομπρέλα προστασίας σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους και την δικαστικέ τις δικαστικές αρχές και τις ανακριτικές αρχές ώστε να μην υπάρχει καμία ανάπτυξη και να μην, ανάμειξη και να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Ε, ευχαριστώ την εισηγήτρια, συνεργαστήκαμε εξαιρετικά. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα πολύ σημαντικό βήμα που κάναμε όλοι από εκεί κοινού. Σας ευχαριστώ πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ ο συνάδελφο Φαντάλεν των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Κάνω μια αναφορά στον κανονισμό. Η κυρία Φώστερ, η αισιόδη συγκήτρια, μου είπε ότι δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα εδώ. Θα καθυστερήσει, θα φτάσει απόψε το βράδυ. Και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το χρόνο αγόρευσή τη. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την συγκήτρια για την εξαιρετική δουλειά τη. Και θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω όλους και όλες που συνέβαλαν στην προετοιμασία αυτού του κειμένου που ασφαλώς θα βελτιώσει τα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλουμε να διδαχθούμε από τα σφάλματα και τα ατυχήματα του παρελθόντος, οι έρευνες πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητες από τις αεροπορικές εταιρείε, από τις οργανώσεις καταναλωτών και κυρίως ανεξάρτητες από τις δικαστικές αρχές. Ως δημόσια υπηρεσία θέλουμε ανεξάρτητες έρευνες. Αυτές όμως οι έρευνες υφίστανται πιέσει. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν ταυτόχρονα να είναι ενδιαφερόμενοι και κριτές και δικαστές. Δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Ε, θα ήταν καλό να είχαμε επιλέξει το καναδικό μοντέλο. Στην Καναδά υπάρχει μια υπηρεσία ανακριτική, τελείως ανεξάρτητη, τελείως αυτόνομη, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και η οποία σε περίπτωση κακοδιαχείριση, σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, ενημερώνει τη δικαιοσύνη. Μία, ένα, υπάρχει επίση στην, στην Ολλανδία ένα ανεξάρτητο ε, σώμα ανακριτών. Κάτι, ένα τέτοιο σύστημα ε, θα ήταν το καλύτερο. γιατί είναι σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία και την αυτονομία της ανάκρισης. Παρόλο που υπάρχουν λήψεις, έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι στο κείμενο. Η υποστήριξη και η προστασία των θυμάτων και των οικογενών τους είναι κατά παραδείγματο χάρη πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Ο κύριος Ζακ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Οι αερομεταφορές είναι οι ασφαλέστερες μεταφορές. Σύμφωνα με τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα, εξίσου εντυπωσιακέ είναι και οι μειώσεις των εκπομπών καυσαερίου. Και θα πρέπει να παραμείνει η κατάσταση αυτή. Η δημιουργία αυτής της υπηρεσίας είναι μια καλή κατάσταση, αλλά θα πρέπει η υπηρεσία αυτή να εξαρτάται από τις δημόσιες αρχές και να μην προσπαθήσει να υποκύψει στην βασική αρχή της άμεσης αποδοτικότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνονται τα πληρώματα των αεροσκαφών στις εταιρείες low cost και πολύ περισσότερα άλλα προβλήματα στα οποία θα πρέπει... Κοιτάξτε, ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν θα πρέπει να περιοριστεί στο να δημοσιεύει ένα μαύρο κατάλογο και να οργανώνει απλά τις ε, έρευνες για, ε, για τα ατυχήματα θα πρέπει να, να ελέγξει τις αεροπορικές επιχειρήσεις και να τις χτυπήσει όταν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πολλές φορές τα ατυχήματα οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε πολλές αεροπορικές επιχειρήσεις, σε επίπεδο εργονομίας, σε επίπεδο κατάρτισης και σε επίπεδο συνθήκων εργασίας. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Αν μιλάτε συνάδελφοι πάρα πολύ γρήγορα δεν είναι καθόλου εύκολο να υπάρξει επαρκής διευμηνία στις υπόλοιπες γλώσσες. Γι' αυτό σας παρακαλώ να μιλάτε λίγο πιο σιγά, λίγο πιο αργά μάλλον, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα από αυτή την πλευρά. Το ίδιο πρόβλημα ε, νιώθω και εγώ εδώ και αρκετά χρόνια. Λοιπόν, περνάμε τώρα στους υπόλοιπους ομιλητές. Ο Ντεγκράντες Πασχουάλ, ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, συγχαίρω την κυρία Ντεβεϊράκη για τη δουλειά που έκανε, που επέτρεψε μια ε, ε, τελική ανάγνωση. Παρ' όλα αυτά θέλω να κάνω κάποιες ε, κριτικές παρατηρήσεις που αφορούν το θέμα της ε, επίτευξης συμφωνίας σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Το πρώτο θέμα είναι το ότι αφήσαμε να μην ε, συμπεριλαμβάνεται το θέμα της ε, ταυτοποίησης των θυμάτων και όχι μόνο σε σχέση με το σώμα των θανόντων και επίσης και για τους συνδέχοντες λόγους και θα υπάρξουν ε, πολλές ε, προσφυγές ε, και είναι σφάλμα εδώ το να υπάρχει μια τεχνική και μια δικαστική διαχωριστική γραμμή. Και εν τέλει η Ισπανική Αντιπροσωπεία θα πρέπει να απόσχει σε σχέση με την θέση που είχε υιοθετήσει υπέρ του θέματος. Και αυτό απλά επειδή από το 1987 βρισκόταν, αντανακλώταν σε σχέση με το αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ το πρόβλημα αυτό και τώρα σε σχέση με το αεροδρόμιο της Κόρτοβα του 2006 προηγούμενες σε σχέση με τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισπανίας και τώρα λόγω μιας αναφοράς επιπλέον. Και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να οδηγηθούμε σε αποχή. Παρ' όλα αυτά είμαστε θετικοί υπέρ της έκθεσης και υπέρ της εργασίας της κυρίας Ντεβεράκα και είναι πραγματικά θετικό το περιεχόμενο της έκθεσής της και αυτό είναι θετικό γεγονός. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Ο επόμενος αγορητής θα είναι ο κύριος Γιάννους Ζέμκε για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα εγώ να πω από πλευράς μου, να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι πραγματικά ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι όλο και καλύτερες επιδόσεις έχουμε στο πεδίο της ασφάλειας στην Ευρώπη. Υπάρχουν ατυχήματα, αλλά γενικά τα επίπεδα ασφάλειας έχουν αναβαθμιστεί και είναι ιδιαίτερα υψηλά. Ωστόσο δυστυχώς η ασφάλεια δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί συλλήβδιν και εξάπαντος διαμιάς. Από καιρού καιρών υπάρχουν ατυχήματα και τέτοιου είδους συμβάντα. Και αυτά, <clears throat> αυτά τα συμβάντα θα πρέπει να εξετάζονται πάντα από ανεξάρτητους ερευνητές επαγγελματικά με πνεύμα επαγγελματικό και ε, με ιδιαίτερη φροντίδα. Αυτό πρέπει να γίνεται ώστε να μπορούν να διατυπώνονται συστάσεις ε, με βάση τα πορίσματα αυτών των ε, ε, ειδημόνων, των ειδικών, ώστε να αποφύγουμε μελλοντικά ατυχήματα και συμβάντα. Σε σχέση με τα όσα υπάρχουν ως διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να μην είναι τόσο καλά όσο θα έπρεπε να ήταν. Υπάρχει δυνατότητα βελτιώσεων λοιπόν. Μέσα στο πλαίσιο της δουλειάς που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλα αυτά μπορούν λοιπόν να βελτιωθούν και να οδηγήσουμε σε βελτιώσεις. Έχουμε λοιπόν ένα εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης στα χέρια μας, το οποίο συνέταξε η κυρία Ντεβεράκα. Ωστόσο όμως από την άλλη πλευρά θα ήθελα να αναφερθώ στα εξής σημεία. Κάποιες παρατηρήσεις και κάποιες τροπολογίες έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση, που είναι το προϊόν συμβιβασμών Πιστεύω ότι θα έπρεπε να ψηφίσουμε επ' αυτόν που ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου. Υπάρχουν άλλες τροπολογίες που θα μπορούσαν να είναι καλοδεχούμενες για κάποιους, θα έπρεπε όμως να απορριφθούν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζέμκε. λέει ο πρόεδρος, ο επόμενος αγορητής η κυρία Μάισνερ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ σε ένα σημείο που ο κύριος Σκιώδης εισηγητής Γέλκο Κάτσιν δεν μπόρεσε για λόγους χρόνου να καλύψει που είναι όμως πολύ σημαντικό. Δεν πρόκειται για την εξέταση των αιτίων ατυχημάτων αλλά για την προστασία των θυμάτων. Και η δική μου κοινοβουλευτική ομάδα άσκησε το επιχείρημα ότι θα πρέπει οι οικοί άμεσα να πληροφορούνται για το τι συνέβη σε σχέση με ένα ατύχημα και να μπορούν να τους συνδράμουν άμεσα. Συνολικά είπαμε ότι πρόκειται για μια πρωτοπόρο έκθεση αυτή που συντάχθηκε από την εισηγήτρια κυρία Ντεβεράκ. Δεν μπορούμε να την επενέσουμε αρκετά. Είναι 16 ετών η οδηγία από το 1994 και χρειαζόμαστε για να εξετάσουμε τέτοια ατυχήματα και συμβάντα με όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούν ε, ανεξάρτητα να διακριβωθούν. Στη ΣΥΠΑ υπάρχουν και ανεξάρτητοι δήμονες ε, και επανείοντες που δρούν ε, ως διερευνητές και αυτό το καταφέραμε τώρα να το πετύχουμε και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Ντεβεράκ για μια εξαιρετική δουλειά που έκανε. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κυρία. Κύριος Μαρινέσκου, παρακαλώ, 1,5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αύξηση, διαρκής αύξηση των εναέριων μεταφορών οδήγησε στην ανάγκη προσαρμογής ε, του νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση ατυχημάτων. Η κυρία Ντεβεράκ πέτυχε ένα εξαιρετικό συμβιβασμό. Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο υπηρεσιών που ασχολούνται με την διερεύνηση ατυχημάτων, με τις βέλτιστες πρακτικές και μια μεθοδολογία που θα είναι κατάλληλη να υιοθετείται από τις ευρωπαϊκές αρχές και να έχουμε καλύτερους μηχανισμού ε, ερευνών και μεγαλύτερη ασφάλεια στις ενέργειες μεταφορέ. Δημιουργήθηκε το αναγκαίο νομικό πλαίσιο για την συμμετοχή της ΕΑΣΑ, ε, του Οργανισμού Ασφάλειας των ε, ε, αναέρων μεταφορών. Και ε, επίσης υπάρχει εδώ και η συμμετοχή ή, και η διαχωριστική γραμμή σε σχέση με τις δικαστικές αρχές και τις ανακριτικές αρχές, ώστε να μπορούν να συντονίζονται, να συντονίστε το έργο, να συντονίστε με το βέλτιστο τρόπο. Η συνδρομή σε σχέση με τους οικείους ε, των θυμάτων από πλευράς των κρατών μελών πρέπει να υπάρχουν προγράμματα και σχέδια ώστε να αντιμετωπίζεται αυτή η ανάγκη. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες και πληροφορίες που θα μπορούν να αναλύονται ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας σε αέριες μεταφορές. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ο κύριος Higgins παρακαλώ στη συνέχεια. Είναι σαφές ότι η προηγούμενη οδηγία έχει πλέον ξεπεραστεί έχει υπάρξει μια έκρηξη στις μεταφορών και χρειάζονται, αερομεταφορών συγγνώμη, και χρειάζεται περισσότερο συντονισμό, περισσότερα μέτρα, περισσότερες επιθεωρήσεις και περισσότερα συνεργασία. Η συγκεκριμένη έκθεση ξεκαθαρίζει τον ρόλο των υπευθύνων αρχών. Υποστηρίζω την πρόταση στην οποία αναφέρθηκε ο Μπράιν Σίμψον και η συγγήτρια ότι η υπηρεσία αυτή σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η ίδια να αναλαμβάνει τέτοιου είδους έρευνες. Ε, θα πρέπει να πιστοποιεί τα αεροπλάνα και τις εταιρείες, αλλά όχι ε, να αναλαμβάνει έρευνες για τα ατυχήματα. Επίσης έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία τα μέτρα για την κατάρτιση των υπευθύνων για τις ανακρίσεις και τις έρευνες ε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται από τα διαφορετικά στάνταρ που επικρατούν στις διάφορες χώρες ο κατάλογο των επιβατών ένα τραγικό στοιχείο λόγω τη καθυστέρηση για τη δημοσίευσή του θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επίση. και η πρόταση έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να δίδεται ένα όνομα επαφής για κάποιον ο οποίος μπορεί να χαθεί σε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια ήδη της κράτησης ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον. Και το θέμα της έρευνας μέσω του DNA. Εν πάση περιπτώσει είναι σωστές οι προτάσεις αυτές. Συγχαίρω την εισηγήτρια και τους χειώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ζασάντα. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Σήμερα συζητάμε ένα έγγραφο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για 800 εκατομμύρια επιβάτες που ταξιδεύουν αεροπορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέτος. Για 16 χρόνια είχαμε έναν κανονισμό ο οποίος είχε ε, αποφασιστεί όταν τότε ε, υπήρχαν πολύ λιγότερες αερομεταφορές. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε τα κατάλληλα επίπεδα ασφαλείας αν δεν έχουμε συγκεκριμένες εθελοντικές παρουσιάσεις και εκθέσεις από πλευρά των πιλότων, των κυβερνητών ε, και των ε, ε, μελών του πληρώματος. Θα πρέπει να νιώθουν ασφαλή όταν αναφέρονται σε συμβάντα τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους δεν θα έχουμε τα κατάλληλα επίπεδα ασφαλείας όταν οι ανακριτικές αρχές και οι ερευνητικές αρχές πιέζονται από τις δικαστικές αρχές, από τις αρχές καταστολής γενικότερα και από τα μέσα ενημέρωσης. Ο καθένας θα πρέπει δηλαδή να μπορεί να κάνει τη δουλειά του με τον κατάλληλο τρόπο. Η ασφάλεια είναι η κορυφή της φροντίδας την οποία θα πρέπει να επιδείξουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ασφάλεια των επιβατών. και οι κανόνες οι οποίοι διασφαλίζουν ε, την ασφάλεια των επιβατών είναι γραμμένοι με το αίμα των θυμάτων των αεροπορικών καταστροφών. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye και έχουμε πέντε που έχουν ζητήσει να παρέμουν. Πρώτος αγορητής, ο κύριος Σαντόβερ, παρακαλώ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια και ένας μήνας από το ατύχημα που άφησε 154 θύματα στο αεροδρόμιο Μπαράχας της Μαδρίτης και πολλών οικογενειών που ε, είχαν ε, ε, θύματα ή κυρίως από τις Κανάριες νήσους. Σήμερα δυστυχώς δύο χρόνια μετά η τεχνική διερεύνηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι οικογένειες των θυμάτων εξακολουθούν να διαρωτώνται τι συνέβη και δεν έχουν απαντήσεις. Και αυτό για δύο λόγους κυρίως. Πρώτα απ' όλα επειδή οι οικογένειες των θυμάτων δεν να αξίζουν να τύχουν τέτοια αντιμετώπιση. Δεύτερον, δεν αποκαλύπτονται θεμελιώδη στοιχεία τα οποία θα ήταν θεμελιώδη σημασία για την ασφάλεια των εναέριων μεταφορών, για την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων. Ομολογώ ότι μεταξύ άλλων αυτή η έκθεση που θα ψηφίσουμε θα διευκολύνει τέτοιου είδου καταστάσει και δεν θα έχουμε τέτοιε επαναλήψει τέτοιων καταστάσεων στο μέλλον. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια που κατάφερε σε πρώτη ανάγνωση να πετύχει μια τέτοια συμφωνία. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να έχουμε τέτοιου είδου συμβάντα για να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκε των θυμάτων. Ο κύριο Λάιχτφιτ στη συνέχεια, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το χειρότερο το οποίο μπορεί να συμβεί, πιστεύω, είναι να είναι κανείς οικείος ενός επιβάτη, γυναίκας ή άνδρα, που έχει αναχωρήσει και μετά να ακούει ως οικείος ότι έπεσε το αεροπλάνο και δεν ξέρουμε ποια είναι η, ε, τι συνέβη με τους επιβάτες. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Εδώ θα ήθελα να πω ότι αυτή η έκθεση είναι κάτι, μια έκθεση που δίνει μια δυνατότητα να μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει επαφή και να συνδρομή όσον αφορά τους οικείους των θυμάτων και να μπορούν ε, να, ε, να διασφαλιστούν οι ανάγκες της συνδρομής. Και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η αβεβαιότητα και ανασφάλεια όταν δεν ξέρουν οι οικοί τι συνέβη ακριβώς και πρέπει να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν αυτή την αβεβαιότητα. Δεύτερον, δημιουργείται μια εξισορρόπηση των συστημάτων εξωτερικών ερευνών και εσωτερικών ερευνών. Είναι πολύ λεπτή αυτή η ισορροπία και πρέπει να πούμε ότι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να ε, καλύπτουν τις ανάγκες μιας ε, έρευνας, από την άλλη όμως πλευρά και εκείνων που πρέπει να καλύψουν ε, τα, τις ανάγκες ασφάλειας στις ενέργειες μεταφορές. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια που κατάφερε να πετύχει αυτή τη σωστή ισορροπία με την έκθεσή της. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Πρόεδρος. Τώρα στη συνέχεια η κυρία Μπιλπάου θα λέει τον λόγο, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμμερίζομαι ότι ο μόνος στόχος αυτού του κανονισμού είναι η πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων σε σχέση με την αποσαφήνιση των ευθυνών. Και χαίρομαι που διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ερευνητών και υπάρχει και η διασφάλιση αυτού του δικτύου ερευνών. Και υπάρχουν διάφορα μέτρα για τα θύματα και για τους οικείους. Προστατεύεται η ευαίσθητη πληροφόρηση, υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας και που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία για άλλους σκοπούς. Κάνουμε λόγους για μητρό, αλλά πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη την αρχή της γιους κουλτούρε, δηλαδή την αρχή της, του σεβασμού της παράδοσης όσον αφορά την προστασία τέτοιων στοιχείων. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το τι πρέπει να κάνουν οι εταιρείε εναέριων μεταφορών ώστε να συνδράμουν τους οικείους των θυμάτων, πράγμα το οποίο δεν διασφαλίζεται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Κυρία Βέτμα, στη συνέχεια παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι ενέργειες μεταφορές διαρκώς αυξάνονται. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα και γι' αυτό πρέπει να έχουμε κάποια ανεξάρτητη αρχή ώστε να μπορεί με ανεξάρτητη δράση να διασφαλίζει το τι πρέπει να γίνει και να υπάρξει η διασφάλιση σε ύψιστο, σε ανώτατο επίπεδο της ε, ασφάλειας. Και γι' αυτό είμαστε υπέρ αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ και σας. Λαν παρακαλώ στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε οι ενέργειες μεταφορές παίρνουν ένα θεμελιώδη ρόλο στην κινητικότητα των ατόμων και στη δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας που καθορίζεται όλο και περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση. Η σημερινή, ε, το σημερινό νομικό πλαίσιο σε σχέση με τέτοιου είδους συμβάντα είναι ξεπερασμένο και εδώ έχουμε και την εμφάνιση νέων ε, εμπλεκόμενων όπως και την, ε, τον Οργανισμό Ασφάλειας των Εναέριων Μεταφορών. Πρέπει να διασφαλίσουμε το ανώτατο επίπεδο από πλευρά των κρατών μελών. Όμω η προτεραιότητα πρέπει να είναι η πρόληψη των ατυχημάτων και η έρευνα πρέπει να είναι βοήθεια πάντα στην πρόληψη. Σημειώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση για τη μείωση του κόστου και αυτό οδηγεί σε αυξημένου κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια. Όμω η οικονομία δεν μπορεί να έχει πριτανεύοντα ρόλο, να είναι πάνω από όλε τι άλλε αρχέ ε, σε σχέση με τη ζωή των ανθρώπων ε, και να δούμε το θέμα των ε, επιβατών Έρευνα ναι, αλλά πρόληψη είναι το πιο σημαντικό και πρόληψη υπέρ των ε, επιβατών. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια εσείς παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ την κυρία Ντεβεράκ για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση για την έρευνα, διερεύνηση και την πρόληψη των ατυχημάτων ε, στην πολιτική αεροπορία θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στις ενεργέ μεταφορές θα έχουν ένα πρόγραμμα υποστήριξης των ε, οικείων των θυμάτων μέσα σε μια προθεσμία δύο ωρών κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να διασφαλίζεται ο κατάλογος των ονομάτων των ε, ατόμων που συμμετείχαν σε μια τέτοια πτήση και θα ήθελα να πω επίσης ότι χαιρετίζουμε την πρόταση να υποχρεούνται εκείνοι οι οποίοι εργάζονται σε αερίες μεταφορές ότι θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις ε, της ε, συμφωνίας ε, του Μορεάλ ακόμα και όταν ένα κράτος δεν έχει επικυρώσει αυτή τη συμφωνία για να αντιμετωπίσουμε με την σωστή πρόληψη τα ατυχήματα και να αποφύγουμε να συμβούν στο μέλλον πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνίες για τις εναέριες μεταφορές με τα κράτη-μέλη. Τελευταίος αγορητής παρακαλώ θα είσαστε εσείς για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πρέπει εδώ να σας αναφέρω, κυρία Πρόεδρε, ότι αν επιτρέπετε, θα ήθελα να προσθέσω ένα στοιχείο που δεν μπόρεσα να αναφέρω προηγούμενα κατά τη διάρκεια του χρόνου της παρέμβασής μου. Η ενημέρωση των οικείων. Οι οικοί πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα. Δεν πρέπει να ασκείται αρνητική μεταχείριση βάρος τους. Όμως η κατάσταση είναι διαφορετική από κράτος σε κράτος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να προστατέψει τα δικαιώματα και τα προνόμια εκείνων των ατόμων που σε κάποιες χώρες αναγνωρίζονται, σε άλλες όμω χώρε δεν αναγνωρίζονται. Υποστηρίζουμε τον ορισμό του τι εστί οικογένεια και πώς θα χρησιμοποιείται αυτός ο ορισμός ε, για την οικογένεια των ε, ε, οικείων, δηλαδή των θυμάτων. Αυτό είναι ένας καλό συμβιβασμός. Το δεύτερο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι σε σχέση με νέους θεσμούς βασιζόμαστε σε ένα δίκτυο αρχών που συνεργάζονται η μία με την άλλη. Τώρα θα λάβει τον λόγο η Επιτροπή παρακαλώ και πάλι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο και δυνατό το μήνυμα προς τα θύματα και τους επιβάτες και τις οικογένειές του. Και αυτό δείχνει ότι έκαναν θαυμάσια δουλειά οι συγγήτρια και οι σχεώδεις συγγητές. Προσβλέπω ε, στο έργο που μας περιμένει για να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα διότι με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουμε την ε, ασφάλεια και την ανεξαρτησία των ερευνών με βάση ε, αποτελεσματική κατάρτιση και υψηλά πρότυπα. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια στις αεροπορικές ε, μετακινήσεις χάρη στην εμπειρία του ΟΑΣΑ του Οργανισμού Ασφάλειας Αεροπορία και θα ήθελα να υπογραμμίσω, όπως είπαν και άλλοι ομιλητέ, ότι θα συμμετέχει ο ΕΑΣΑ ω σύμβουλο τεχνικός για να μοιραστεί την εμπειρία και τις γνώσεις του με τους, ε, τις υπηρεσίες χωρί χωρίς να αναλαμβάνει ο ίδιος ανακρίσεις. Εμείς θα, θα, επιταχύνουμε τη διαδικασία εξυγχρονισμού, εξυγχρονισμού των διατάξεων, ώστε τελικά να έχουμε τα καλύτερα μέσα στη διάθεσή μας για να κάνουμε σωστή δουλειά προστατεύοντας τη ζωή των Ευρωπαίων επιβατών και ταξιδιωτών. Σας συγχαίρω και πάλι για το έργο σας. Ευχαριστούμε θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα λάβει τώρα εκ νέου τον λόγο η κυρία Ντεβεράκ Ευχαριστώ για τη συμβολή σας και όλους και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία διευκόλυνε σημαντικά το έργο μας. Θέλω να καθυσυχάσω τον κύριο Ζέμκε. Αύριο θα υπάρξει μόνο μία τροπολογία. Πρόκειται για ένα λάθο. Το Συμβούλιο είχε ξεχάσει μία παράγραφο στο κείμενο. Αναζητήσαμε τον καλύτερο τρόπο να το εντάξουμε και πάλι αυτή την παράγραφο στο κείμενο μέσω μια τροπολογία, μοναδική τροπολογία. Ο κύριο Χίγκιν ίσω δεν με άκουσε για τόση πολύ φασαρία όταν ξεκίνησα την ομιλία μου και το επανέλαβε η κυρία Μάλστρομ ότι ο οργανισμό που θα παίζει θα έχει ρόλο πιστοποίηση δεν μπορεί να αναλαμβάνει την έρευνα, τη διερεύνηση των ατυχημάτων, αλλά θα έχει πρόσβαση σε όλα τα αναγκαία στοιχεία για να ασκήσει το, για να ε, ε, ασκήσει το ρόλο του ως αρχή πιστοποίησης συνδράμοντας και υποστηρίζοντας το ανακριτικό έργο. Το, αυτό που καταγγείλατε νομίζω ότι βελτιώθηκε, δηλαδή την έλλειψη πληροφοριών, η αβεβαιότητα των οικογενειών. Στην πρώτη ανάγνωση οι σκιώδεις ηγητές θα σας πούν αυτό που λέω και εγώ ότι το κοινοβούλιο δεν υποχώρησε, υποχώρησε σε τίποτε στην πρώτη ανάγνωση. Επικράτησαν σε όλα τα θέματα του κειμένου οι απόψεις του κοινοβουλίου. Είμαι πολύ ευτυχής που το κείμενο αυτό που όπως είπε ο Κιούνα αναφέρεται ε, αφορά ε, ανθρώπινες ζωές ε, εξασφάλισε τη συνένεση των πολιτικών ομάδων. Νομίζω θα υπάρξει μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης αύριο ώστε να επιβεβαιώσουμε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως κινητήρια δύναμη για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών τους, ώστε να μπορούν να ζουν σε μια Ευρώπη που πραγματικά φροντίζει για την ασφάλειά τους. Σας ευχαριστούμε θερμά. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε τώρα. Η ψήφιση θα γίνει αύριο το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι. Η ψήφιση της έκθεσης. Αξιότιμοι συνάδελφοι, επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη.